Επίσης, μαζί με το Πρόεδρο του Συμβουλίου όλες τις πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 78 του κανονισμού του Κοινοβουλίου. Τα, οι τίτλοι θα δημοσιευθούν στα πρακτικά αυτής της συνόδου.